της τον Οκτώβριο. Λοιπόν, βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης επιγράφεται το βραβείο. Τιμά με μονομένα πρόσωπα, προσωπικότητες ή και ε, οργανώσεις που με θάρρος υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και γενικά με μεγάλη ευθύνη ζουν πάρα πολύ επικίνδυνα στον αγώνα τους κατά της μυσαλλοδοξίας και της καταστολής. Έχει αποκτήσει κάποια έγκλη πλέον το βραβείο, γνωρίζετε ποιοι έχουν τιμηθεί. Εξαιρετικές προσωπικότητες που καταπολεμούν τη μυσαλλοδοξία και το φανατισμό. Και το πιο εύκολο το παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Ανδρέης Ζαχάροφ, του οποίου το όνομα φέρει το έγγραφο. 60 χρόνια αγωνίστηκε με εξαιρετικό θάρρος και το πλήρωσε και πικρά. Ήταν ε, τιμόμενο πρόσωπο, προσωπικότητα ως επιστήμων στη Σοβιετική Ένωση. Και παρόλα αυτά δεν δέχτηκε να βολευτεί αλλά αγωνίστηκε για την ελευθερία της έκφρασης και τα ανθρώπινα δικαιώματα με απίστευτο θάρρος και το πλήρωσε πάρα πολύ πικρά. Και φέτος έχουμε μια σειρά προτάσεων που συζητήσαμε και χαιρόμαστε ε, που λαμβάνει και φέτος χώρα. Το 2008 που ήταν 20 ετία του βραβείου Σαχάροφ, ο τότε πρόεδρος του Κοινοβουλίου, κύριος Πέτερινγκ, δημιούργησε ένα δίκτυο βραβείου Ζαχάροφ που θα αποτελεί μια πλατφόρμα για να μπορούν να έρχονται σε επαφή ε, οι κάτοχοι του βραβείου να επικοινωνούν, να συνεννοούνται με αλληλεγγύη. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτό θα λάβει σάρκα και οστά το Ίδρυμα, πώς θα υπάρχει μόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αυτών των προσωπικότητων και να ε, βοηθήσει έτσι περαιτέρω το κοινό μας ε, στόχο. Σας ε, θυμίζω και σας ενημερώνω στις 10 Οκτωβρίου 4.30 με 5.30 θα υποδεχθούμε τρεις βραβευθέντες του 2011 σε μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών υπό Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για ε, την προσωπία για τις χώρες μα και για την προσωπία για τι χώρες Μακρέπ καθώς επίσης και την Αραβική Ένωση του Μακρέπ. Δεν βλέπω εδώ την Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να ρυθμιστεί κάπω, Δεν ξέρω γιατί δεν συμμετέχει η Επιτροπή Ανάπτυξη, αλλά βεβαίω είναι ευπρόσδεκτοι και οι συνάδελφοι. Ε, θέλω να δώσω όμω το λόγο στην κυρία Στριφλέρ και την Προεδρία, γιατί πρέπει να φύγω και χαίρομαι για την παρουσίαση των υποψηφίων. Mon cher collègue, euh, Monsieur merci. Bonjour, euh, cher collègue. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μπρόκ, κύριοι συνάδελφοι, πριν παρουσιάσω τους υποψηφίους, θα ήθελα να υπενθυμίσω πώς είχαν οι προηγούμενες φάσεις της διαδικασίας. Όταν εξέπνευσε η διορία κατάθεση των υποψηφιωτήτων στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, η γραμματεία είχε λάβει πέντε, προτα... πέντε υποψηφιότητες των σοσιαλιστών, των φιλελευθέρων, των πρασίνων και τα λοιπά. Καθώς και του συναδέλφου Σαλαφράνκα, Έλμαρ Μπρόκ και 11 άλλων. Πριν μιλήσουν οι συνάδελφοι για τους προτιμόμενους υποψήφιους θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει πάνω από 5 λεπτά ακόμη και αν πρόκειται για συλλογική υποψηφιότητα. Θα επιμείνω ιδιαίτερα σε αυτόν τον κανόνα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο πόσο μάλλον που είναι πολλοί υποψήφοι και θέλουν να τους παρουσιάσουν πολλοί συνάδελφοι. Ορισμένες παρουσιάσεις μπορούν να συνοδεύονται και από ένα σύντομο φίδεο ή από διαφάνειες. Η γραμματεία έλαβε ταινιούλες για τον υποψήφιο κύριο Ιωσήφ Φράγκης. Θα αρχίσει λοιπόν τώρα η παρουσίαση των υποψηφίων από τους σπόνσορές τους και οι τελευταίοι αυτοί θα μας πούν σύντομα τι έχουν καταφέρει οι υποψήφοι για την ελευθερία του πνεύματος. Καταρχήν λοιπόν θα δώσω το λόγο στο συνάδελφό μας Γιάτσεκ Σαριούς Βόλσκι για να μας παρουσιάσει τον κύριο Αλές Μπιαλάτσκι που βρίσκεται φυλακισμένο στη Λευκορωσία. Έχετε το λόγο για πέντε ολόκληρα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν είναι πρόταση πολιτικής ομάδας, αλλά μιας διακομματικής ομάδας ευρωβουλευτών, γιατί τέτοιος είναι και ο υποψήφιος. Εκπροσωπεί τις αξίες που όλοι συμμεριζόμαστε εδώ μέσα, χωρίς κομματικές, κομματικούς φραγμούς. Είναι μαχητής της ελευθερίας από τη Λευκορωσία, ευρωπαϊκή χώρα και γειτονική μας, που έχει υποστεί καταπίεση και δικτατορία με πολύ γνωστότερους τρόπους. Μέχρι τώρα η Ένωση και το Κοινοβούλιο μας λίγα έχει πράξει για την υπέρ της Λευκορωσίας και είναι εδώ ευκαιρία να κάνουμε κάτι παραπάνω για να δώσουμε το μήνυμα στη Λευκορωσία ότι δεν ξεχνάμε τον αγώνα όσων αγωνίζονται και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Σήμερα εξάλλου είναι και τα γενέθλια του Άλες Μπιαλάτκι που θα τα γιορτάσει στη φυλακή είναι ο άνθρωπος που έχει φυλακιστεί για τον περισσότερο χρόνο επί του τωρινού Προέδρου Λουκάσενκο. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο πιστεύω του ίδιου του Σάχαροφ. Πρόκειται δηλαδή για άνθρωπο που δεν λύγησε ποτέ στον αγώνα του χωρίς να σκέφτεται το τίμημα είναι σημαντικό λοιπόν να τον προστατεύσουμε δίνοντάς του αυτό το βραβείο γιατί αυτό νομίζω θα τον βοηθούσε στους επόμενους αγώνες του. Μερικοί λένε ότι έχει δοθεί και σε άλλον Λευκορώσο το βραβείο, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους γεωγραφικές κατανομές και ποσοστώσεις στατιστικά εξάλλου. Τρία βραβεία πήραν η Κούβα και τρία το Κωσυφοπέδιο, δύο η Κίνα, η Συρία και η Νευκορωσία και από τα 33 βραβεία που έχουν συνολικά δοθεί μόνο 9 δόθηκαν σε Ευρωπαίους. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε τι συμβαίνει και στις γειτονικέ μας χώρες. Ο Άλες Μπιαλάτσκι υποστηρι... υπολογίζει στην υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρέδα για να μας πει για ποιους λόγους αυτός και άλλα μέλη της ομάδας του υποστηρίζουν την διπλή υποψηφιότητα που υποστηρίζουν. Όχι! Θα λάβουμε το λόγο, αλλά για μια άλλη υποψηφιότητα των δύο Ιρανών Μπορώ να το κάνω τώρα, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαρίστω. Ναι, αλλά εδώ φαίνεται υπάρχει τεχνικό πρόβλημα που λέμε. Δεν έχω τα σωστά τετράδια εδώ μπροστά μου. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Τάνοκ τώρα για να μας παρουσιάσει την υποψηφιότητα που υποστηρίζει αυτός και η ομάδα του και ο κύριος Πέτερμαν. Επίσης ε, τον κύριο Γιώζεφ Φράνσις του Πακιστάν. Αλλά μαζί να μην ξεπεράσουν τα πέντε λεπτά. Κύριε Πρέντα, συγγνώμη, αλλά να. ευχαριστώ. Το θέμα το πρόσωπο που προτείνουμε είναι ο κύριος Ιώζεφ Φράνσις από το Πακιστάν. Έχετε ακούσει εσείς για τον νόμο περί βλασφημίας στο Πακιστάν. Έχουν υπάρξει συζητήσεις και ψηφίσματα γι' αυτό τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ορισμένε ε, ε, νομικές ρυθμίσεις. Ε, είναι οι ρήτρε χατούν της Σαρία, του νόμου του Ισλαμικού που οδηγεί στην φυλάκιση και στην θανάτωση, στην εκτέλεση αυτών για τους οποίους υπάρχουν ε, υποψίες και όσοι καταδικαστούν έτσι και αλλιώς με, σύμφωνα με αυτούς τους νόμους κινδυνεύουν να πεθάνουν και από τις ε, άτακτες μορφές χειροδικίας. Ε, χρησιμοποιούνται οι νομικές αυτές ρυθμίσεις και για, την, ε, για προσωπικούς λόγους εις βάρος ορισμένων προσωπικών εχθρών και πρόσφατα έχουμε το παράδειγμα ενός κοριτσιού 14 ετών που κατηγορήθηκε για βλασφημία εναντίον ε, των γειτόνων της από ένα ημάμι, αλλά ευτυχώς από ό,τι φαίνεται η εισαγγελία την αθώωσε. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια θύματα, χριστιανοί και μουσουλμάνοι οι συνέπειες αυτές δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα αυτή η οποία υποφέρει από ένδυα, εξτρεμισμό και τα παιχνίδια εξουσίας. Είχαμε ένα ψήφισμα και για τη δολοφονία του κυβερνήτη του Πουντζάμπ, όπως επίσης και του Υπουργού του Χριστιανού που δολοφονήθηκε επειδή άσκησαν κριτική στους νόμους αυτούς βίες διαδηλώσεις προκαλούνται από περιπτώσεις βλασφημίας τους τελευταίους μήνες. Ο υποψήφιος λοιπόν, ο Γιώζεφ Φράνσις, είναι ένας από τους λίγους πια, οι οποίοι με μετριοπαθή τρόπο αμφισβητούν τους νόμους περί βλασφημίας και τους αμφισβητούν λόγω των καταχρήσεων που προκαλούν. Ε, και σε τη άλλη θυμίζω ότι από την Νότια Ασία τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε κανένα υποψήφιο και πρέπει να μην αγνοούμε το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή του πλανήτη, ιδιαίτερα στο Πακιστάν, όπου θεωρητικά τουλάχιστον είναι δημοκρατία, υπερασπίζεται τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες με τη Δύση, αλλά δυστυχώς αυτοί οι νόμοι αμφισβητούν αυτή τη διαπίστωση. Ο Πέτε Βαντάλεν θα σας παρουσιάσει τώρα την προσωπικότητα του Ιώζεφ Φράνσις. Ευχαριστώ πολύ, Φέτος υποστηρίζουμε τον Γιώργο Φράνσις και ελπίζουμε ε, τον Οκτώβριο να μας βοηθήσετε ε, για να περάσει αυτή η υποψηφιότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το 1992 ο Γιώζερ Φράνσις ίδρυσε το Κέντρο για την Νομική Συνδρομή και τους διαγνωνισμούς. Ε, εκεί απευθύνονται θύματα της νομοθεσίας περί βλασφημίας στο Πακιστάν και η δουλειά αυτής της οργάνωσης είναι να υποστηρίζει τα τυχόν θύματα με δεκάδες ε, δικηγόρων που παρέχουν ε, δικαστική, νομική μάλλον συνδρομή ε, και η κυρία Μπίμπη είναι ένα από τα θύματα που ήρθε στα γραφεία για να ευχαριστήσει την οργάνωση για την αθώωσή της μαζί με το σύζυγό της. Αυτό το κέντρο επίσης φροντίζει να υπάρχουν και ασφαλείς ε, κατοικίες ή στέγη για εκείνους που διώκονται για βλασφημία και τους ε, υποστηρίζει με τρόφιμα και χρήματα. Σε άλλη φωτογραφία βλέπετε ε, τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Ζωζε Φράνσις κατά της νομοθεσίας αυτής στο Πακιστάν και ζητάει την ανάκληση αυτών των νόμων. Και η τελευταία φωτογραφία σας δείχνει ε, την επίσκεψη του Ζόζεφ Φράνσις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήρθε αρχές το έτος για να μας εξηγήσει πώς έχει κατάσταση στο Πακιστάν και τι ισχύει με την νομοθεσία περί βλασφημίας. Και τότε που συμφώνησε για την υποψηφιότητά του. Πραγματικά σας απευθύνουμε έκκληση, σας συγκετεύουμε να τον υποστηρίξετε. Επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο περάσαμε ψηφίσματα κατά της νομοθεσίας παρήβλασφημίας και αν τον υποστηρίξουμε θα δείξουμε ότι... Η ανεξιθρησκεία, η ελευθερία της έκφρασης είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και η κατάσταση στο Πακιστάν, ιδιαίτερα για ανθρώπους όπως ο Ζουζερ Φράνσις που ε, έχει ε, αφιερώσει τη ζωή του ολόκληρη σε αυτόν τον καλό σκοπό. Γι' αυτό σας ε, ζητούμε να υποστηρίξετε αυτόν τον τόσο αξιόλογο υποψήφιο. Ευχαριστούμε πολύ. Merci beaucoup. Donc, euh, nous Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον Σαντιάγο Φίσας και στον Βίλι Μέγερ που θα παρουσιάσουν την ομαδική υποψηφιότητα της κυρίας Σομόσα του κυρίου Ταγκαντά, του κυρίου Μουσαϊντή, που είναι αντιπολιτευόμενοι την εξουσία στη Ρουάντα στο Κιγκάλι. Παρακαλώ και οι δύο να μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά. Ο κύριος Φίσας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας αγαπητοί ε, συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της ε, υποψηφιότητας των τριών εκπροσώπων της ε, αντιπολίτευσης στην. Ε, Ρουάντα, Βικτουάριν Γκαμπίρε, Ντεοκράσια Μουσαΐντι και Μπερνάρν Τανκάντα. Κρατούνται στη χώρα τους, ήταν κατά της βίας και υπέρ της συμφιλίωσης. Έχετε το σύντομο βιογραφικό τους όλοι στα χέρια σας, οπότε δεν θα σας εξηγήσω ε, εκτενώς την κάθε περίπτωση. Απλώς ε, να πω ότι υποστηρίζεται αυτή η υποψηφιότητα από βουλευτές διαφόρων πολιτικών κομμάτων, του Λαϊκού Κόμματος, ε, των Σοσιαλιστών και της Ενωτικής Αριστεράς. Η υποψηφιότητα αυτή μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική, διότι τα τελευταία χρόνια το βραβείο Σαχάροφ επικεντρώνεται σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, Κούβα, αραβικές χώρες, η Λευκορωσία και κάπως είχε παραγωνιστεί η Αφρικανική Ήπειρος, ε, προκειμένου η Ρουάντα. Όπως γνωρίζετε όλοι, η χώρα αυτή ζει μια δικτατορία που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είναι βαθύτατος ο διχασμός εθνοτικός μεταξύ των δύο βασικών φυλών ε, που είναι η Χούτου και η Τούτσι. Οι, υποψήφοι μας αυτοί χρόνια αγωνίζονται για να αλλάξει η κατάσταση και κατέληξαν στη φυλακή όπου υφίστανται τα πάνδυνα. Ε, κακοποίηση και βασανιστήρια. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στη Βικτόρ Ιγκαμπίρε που είναι γυναίκα και ε, μετά ε, την αναγκαστική της εξορία στις κάτω χώρες έφτιαξε οικογένεια και είχε και επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά θέλησε να γυρίσει στη χώρα της για να κάνει κάτι να τη σώσει από τη δικτατορία και να προσπαθήσει να προωθήσει την οδό του διαλόγου μεταξύ των τριών εθνοτήτων Χούτου, Τούτσι και του που είναι η μόνη λύση ο διάλογος πάνω από 1,5 χρόνο κρατείται και δεν έχει επικοινωνήσει με τον άντρα της και τα τρία της παιδιά στην Ολλανδία. Δεν θεωρώ ότι είναι ε, λιγότερο σημαντικές οι άλλες υποψηφιότητες, αλλά πιστεύω ότι αν, ε, το, απονείμουμε το βραβείο τους ε, υποψηφίους από τη Ρουάντα, θα δείξουμε τη σημασία την οποία αποδίδουμε και στη χώρα και στους τρεις αυτούς αντιφρονούντες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ο κύριος Μάγερ. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου Σαντιάγο Φίσας, η Ρώσα Σταρά, η Μαρία Μουνίθ, η Άννα Μιράντα και άλλοι 37 βουλευτέ συνυπογράφουν αυτήν την υποψηφιότητα, όπω ακούσαμε από διάφορε πολιτικέ ομάδε, Πιστεύω ότι έχουμε εδώ μια ευκαιρία να δώσουμε θετική απόκριση σε εκείνου που θέλουν η Ρουάντα να είναι ένα έθνος συμφιλειωμένο για να ε, σταματήσει όλη αυτή η, πολιτική, ε, πολιτιστική αποκλεισμού και βίας στη Ρουάντα. Και οι τρεις είναι πάρα πολύ αφοσιωμένοι στην ιδέα της συμφιλίωσης. Έχουν διαφορετικό βιογραφικό, προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές ε, δυνάμεις. Μάλιστα ο ένας είναι Τούτσι, που τότε είχε καταγγείλει όλη αυτή τη βία απέναντι στους Χούτου και οι τρεις λοιπόν είναι το πιο εύγλωτο παράδειγμα που θα μπορούσε να δώσει κανείς για τη συμφιλίωση. Επίσης θεωρούμε πάρα πολύ σκόπιμο και επίκαιρο να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιταχυνθεί και η διπλωματική οδός για να αφαιθούν ελεύθεροι οι τρεις αυτοί κρατούμενοι και πιστεύω ότι το βραβείο Σαχάροφ είναι ένα βραβείο που τους αξίζει και στους τρεις διότι ανταποκρίνονται σε όλες τις προϋποθέσεις και είναι και σύμβολο για το ποια μπορεί να είναι αυτή η συμφιλειωμένη Ρουάντα. Πιστεύω λοιπόν ότι η πρότασή μας συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να υποστηριχθεί, να προωθηθεί και θα ήταν και ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα για την Αφρική και ε, για ε, το τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία θεωρώ σημαντικό και οι τρεις και η Βικτόρια ο Μουχώσα και ο, ο Τεοκράσιας Μουσαϊντή και ο Μπέρναρ Ταγκάντα να έχουν την ευκαιρία να αφαιθούν ελεύθεροι και να έρθουν να παραλάβουν το βραβείο Σαχάροφ και οι τρεις. Ε, ευχαριστώ. Ωραία. Τώρα ο συνάδελφος Σούλτς των Πρασίνων για να υποστηρίξει τη σπούση Ράιοντ δηλαδή Ναντιέσδα Αντρέγεβα Τολοχονίκοβα, Εκατερίνη Σαμούσεβιτς και την Μαρία Αλιόχινα. Ορίστε κύριε Σούτς μου. Πολύ ωραία τα προφέρετε τα ονόματα, κυρία Πρόεδρε. Αναγνωρίζουμε και έχουμε επίγνωση ότι και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι αξίζουν το βραβείο Ζαχάροφ. Θα ήθελα εγώ να προτείνω το group punk ε, Pussy Riot. Δεν χρειάζεται στη Ρωσία επιπλέον να εξηγήσουμε τι εστί βραβείο Ζαχάροφ, γιατί εκεί χαίρει μεγάλου ηθικού κύρους και ειδικού βάρους. Γιατί εγώ γνώρισα και τον Ανδρέη ε, Ζάχαροφ και τη ε, σύζυγό του Έλενα Μπόραν που πέθανε πρόσφατα. Είμαι βέβαιος ότι θα ήταν στο πλευρό αυτών των θαραλέων κοριτσιών που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του λαού. Ο Σολτζενίτσιν ε, το είπε ε, πολύ εύγλωτα στον πρώτο κύκλο της κολάσεως ότι τα λόγια μπορούν να σπάσουν τον πετόν. Ε, είχαν λοιπόν εσωτερικό σθένος και θάρρος και στράφηκαν κατά αυτού του ε, αυταρχικού καθεστώτος, του πατριαρχικού καθεστώτος, κρατικής βίας με το δεσποτικό χαρακτήρα και τη νομική και δικαστική ε, αυθαιρεσία. Όλα αυτά τα αποκάλυψαν. Το Σεπτέμβριο πέρσι ιδρύθηκε ε, αυτό το γκρουπ με αφορμή αυτή την κοινική αλλαγή φρουρά στην εξουσία Πούτιν Μετβέτιεφ και ήθελαν να καταγγείλουν αυτό το κίνδυνο ότι επιστρέφει η αυταρχική αχείριση στην Ρωσία και μετά ε, την αναβική Άνοιξη διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες είναι και αυτές οι χαμένες των εξελίσσεων. Ε, οι γυναίκες λοιπόν ε, εξεγείρονται και ε, δεν θέλει ούτε να, να προφέρει ε, το όνομα του γκρουπ ο, ο κύριος Πούτιν όπως κατά τα άλλα θα χαρακτηρίζει τις λευκές κορδέλες που φορούν οι γυναίκες και οι διαδηλωτές προφυλακτικά ή θέλει να κρεμάσει τον κύριο Σακασβίλη όπως θα θυμάστε. Ε, λοιπόν δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Είναι ένα κράτος το οποίο... Ε, απέχει και απομακρύνεται από το κράτος ε, δικαίου και τις δυτικές αξίες. Είναι και συμβολικό αυτό ότι έγινε. Να το εξηγήσω για να το καταλάβουμε καλύτερα. Το 1968 δύο νεαρές ε, ε, γυναίκες στην Κόκκινη Πλατεία με πανό διαδήλωναν κατά την εισβολή στην Πράγα και καλοκαίρι ήταν και φορούσαν παλτά για να προετοιμαστούν για τη Σιβηρία γιατί ήξεραν ότι θα τους συλλάβουν. Και ε, ε, φέτος το χειμώνα ήρθαν οι γυναίκε με καλοκαιρινά ρούχα και διαδήλωναν πάλι στην κόκκινη πλατεία κατά του Πούτιν και είπαν ότι δεν θα μα τρομάξετε. Είναι και ένα είδος ε, τέχνης, ε, ο κοσοπτουαλισμός της Μόσχας που είχε καταγγείλει ε, την κατάσταση. Δεν είναι βλασφημία, ήταν μια προσευχή πανκ. Καμία σχέση με βλασφημία. Ε, προσεύχεται στην Παναγία τον γκρουπ να τους λυτρώσει, να τους απελευθερώσει. Όταν ε, ε, ήθελε κανείς να ξεφορτωθεί στους Μπολσεβίκους ή τον Ιβάν τον, τον Δρομερό και άλλους που κατέστραφαν εκκλησίες, στην Παναγία προσεύχοντα. Για να τους σώσει από τον πονηρό. Και τώρα, ο Πούτιν λέει ότι θέλει να προστατεύσει την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους χώρους λατρείας. Ναι, αλλά η ίδια η Εκκλησία ε, έχει ξεχάσει ότι δεν έχει ε, ανατινάξει ο Στάλιν και μάλιστα ε, με ενθουσιασμό των πολιτών. Και πολύ κοντά στη Λιουμπιάνκα πήγαιναν και για μπάνιο διάφοροι και δεν είχαν κανένα πρόβλημα Και εδώ οι γυναίκες αυτές καταγγέλουν τη διαπλοκή μεταξύ του Πούτιν του Τρίτου και του Κυρίλου του Πρώτου και επιτίθενται γιατί δεν θέλουν να γίνει θεοκρατικό κράτος ε, η, Ρωσία όπως το Ιράν, να υπάρχει ορθόδοξος πολιτισμός, γιατί αυτή τη στιγμή η Ρωσία προς τα εκεί οδεύει. Και να διασκεδάσω και μια προκατάληψη. Πολλοί συνάδελφοι λένε ότι εντάξει, σε εμά θα ήταν διοικητικό πρόστιμο, δεν του επιβλήθη πολύ βαριά ποινή, δεν επιτρέπεται αυτό. Μα σε εμά ούτε πρόστιμο. Κανένα group punk ε, δεν χρειάζεται να πάει σε μια εκκλησία και να ζητήσει να φύγει ε, η ηγεσία της χώρας, γιατί έχουμε νόμιμους τρόπους, εξεταστικές επιτροπές, ε, σε κοινοβούλια, διαδηλώσεις. Επειδή είναι αυτό το καθεστώς τόσο αυταρχικό, είναι και ο τρόπος διαμαρτυρίας τόσο ακραίος. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα οι συνάδελφοι Πρέδας, Βερονίκη Ντεκέιζερ, Μαριέτε Σάκε και Ελένη Φλότρ να μας παρουσιάσουν τους δύο Ιρανούς που είναι η κυρία Ναστρίν Σότουντεχ και ο κύριος Τζαφάρ Παναή. Και αυτοί να μην ξεπεράσουν τα πέντε λεπτά που διαθέτουν όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι βέβαια δύσκολο να διαλέξει κανείς, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε όπως και τα προηγούμενα χρόνια να αναζητήσουμε κάποιο συμβιβασμό ή συνένεση. Επειδή είμαστε πολλοί σπόνσορες, θα πω τα γενικά εγώ και μετά οι συνάδελφοι τα ειδικά. Η χώρα είναι χώρα που βρίσκεται στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων όπου η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθε είναι περιορισμένη, είναι χώρα όπου υπάρχουν βασανιστήρια καθημερινά, όπου επιβάλλονται υπερβολικές ποινές. Μετά την Κίνα μάλιστα το Ιράν είναι δεύτερη στις εκτελέσεις ήταν το 2011. 360 άνθρωποι εκτελέστηκαν πέρυσι και κατά υπενθυμίζοντας ότι στη χώρα αυτή υπάρχει ολόκληρη στρατηγική καταπίεσης από το κράτος και δίνω το λόγο στους υπόλοιπους σας κατευχαριστώ. Κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι επίσης και χώρα με μεγάλους καλλιτέχνες και με μεγάλο πολιτισμό και θα ήθελα να πω ότι το καταπιεστικό καθεστώς του Αχμαντίν Τζάντ δεν κατάφερε ποτέ να τους κάνει να σιωπήσουν, να τους φημώσει. Και για τον Τζαφάρ Παναχή που υποστηρίζω μπορώ να σας δείξω και το πρώτο του έργο που έστειλε στις Κάνες το 1995 το άσπρο μπαλόνι. Και ήταν πολύ καλό όπως εξάλλου πολλά ιρανικά έργα. Τώρα, μερικά λόγια για τον Τζαφέρ Παναή. Δεν κάνει πολιτικά έργα, αλλά έργα που μιλούν για την κοινωνική πραγματικότητα. Ήθελε να εκφραστεί γιατί η σιωπή λέει είναι θάνατος. Ο Παναή για μας εκπροσωπεί τον αγώνα κατά της καταπίεσης και αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας έκφρασης. Είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος μεταξύ των σημαντικότερων του Ιρανικού νέου κύματος. Άρχισε από το 69, Μότε Φαϊχβέντ λεγόταν το κίνημα. Τα έργα του Τζαφάρ είναι απαγορευμένα στο Ιράν σήμερα, αν και με μορφή DVD πολλούνται κρυφά. Είναι πολύ γνωστό στο εξωτερικό που έλαβε πολλά βραβεία, ιδιαίτερα στις Κάνες, στο Βερολίνο και στη Βενετία τα έργα του καταδικάζουν την αδικία, τις κοινωνικές ανισότητες και την άνηση μεταχείριση κατά των γυναικών. Ίσως έχετε δει το έργο των Ιρανών γυναικών που πήγαιναν κρυφά να δουν ποδοσφαιρικούς αγώνες γιατί απαγορεύεται στις γυναίκες να μπαίνουν στα γήπεδα από το 79 και μετά. Μετά από την επανεκλογή του Αχμαντινετζάντ, την οποία πολλοί αμφισβήτησαν το 2009, ο Τζαφάρ έκανε ένα ντοκιμαντέρο που έδειχνε τις μαζικές διαδηλώσεις και αυθόρμητες του Ιρανικού λαού που καταπιέστηκαν σκληρά. Και μετά από αυτό το έργο συνελήφθη την 1η Μαρτίου 2010 με 16 άλλους εξώνυγοι τη γυναίκα του και την κόρη του μετά από απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την κακομεταχείριση ε, απελευθερώθηκε με εγγύηση το 2010 τον Μάιο αλλά μετά από λίγους μήνες πάλι συνελήφθη για αντιιρανική δραστηριότητα και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθυρξης και 20 έτη απαγόρευσης κινηματογράφησης. Παρά τις αμαρτυρίες της διεθνούς κοινότητας τον Οκτώβριο του 2011 επιβεβαιώθηκε η καταδίκη του και είναι πάλι ακόμα στη φυλακή. Πράγμα το οποίο δεν τον εμποδίζει να συνεχίζει τον αγώνα του συγγράφοντας μαζί με έναν άλλον το γνωστό έργο «Αυτό δεν είναι έργο» που κάνει μια παραπομπή στο γνωστό πίνακα του Μαγκρίτ το οποίο έργο βγήκε από το Ιράν σε ένα κλειδί USB και παρουσιάστηκε εκτός συναγωνισμού στις Κάνες το 11. Αυτόν το σκηνοθέτη θα θέλαμε να βραβεύσουμε. Θα θυμίζει ίσως η περίπτωσή του και τους σοβιετικούς αντιφρονούντες και για, τον, για την αστρίνσο του Ντε θα μιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Έληξε ο χρόνος ομιλίας, αλλά δεν μπορώ να μην δώσω το λόγο και στους δύο υπόλοιπους. Πρέπει όμως να βιαστούν. Η κυρία Μαριέτσε Σάκε. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Είναι καιρός να πάει σε Ιρανούς το βραβείο Σαχάραφ. Η ρητορική και τα δόγματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έχουν πλέον καμία νομιμοποίηση λαϊκή η καταστολή έχει αυξηθεί και προσπαθούν να σιωπήσουν όλες τις φωνές που ακούγονται και που αμφισβητούν το καθεστώς και ιδιαίτερα τις γυναίκες. Ξέρουμε τι έγινε με την εξέγευση του 2009. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν από το Ιράν. Αυτοί που παρέμειναν δίνουν μάχη με μεγαλύτερο ακόμα θάρρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό η Ναστρίν Σουτουντέ αξίζει να πάρει το βραβείο. Είναι μια εξαιρετική υποψήφιος, ε, είναι δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι φυλακισμένη, έχει υπερασπιστεί νέα παιδιά και κοπέλες οι οποίοι είχαν πέσει θύματα βιοπραγιών στα σπίτια τους. Κοιτάξτε, έχετε ξεπεράσει τον χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας, που είχαν οι προηγούμενοι ε, υποψήφοι Κοιτάξτε, όλοι οι υποψήφοι είναι ενδιαφέροντες. Κοιτάξτε, ούτε μισό λεπτό δεν μίλησα, λέει η κυρία Σάκε. Είναι γελίο, λέει η κυρία Σάκε, αυτό το μέτρο που εφαρμόζεται. Όλος ο χρόνος για όλου, ε, όλους, παρακαλώ, για την παρουσίαση των υποψηφίων υπάρχουν κανόνες. Κυρία Φλότρο, θέλετε να τελειώσει η κυρία Σάκε. Κοιτάξτε, δεν είμαστε μηχανές. Οι κανόνες είναι κανόνες, λέει η κυρία Στρίφλερ. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να ερμηνεύσετε τους κανόνες και τους ερμηνεύετε όπως σας καπνίσει, λέει η κυρία Σάκε. Κοιτάξτε, λέει η κυρία Στρίφλερ, μου ζήτησα να είμαι αυστηρή ή είμαι αυστηρή. Και σέβομαι τους κανόνες, καλό θα ήταν να τους σέβονται όλοι. Κοιτάξτε, 15 δευτερόλεπτα μου δίνετε, οπότε λέει η κυρία Φλότρο θα πω το εξή. Ανάμεσα σε όλους που πήραν το βραβείο Σαχάροφ, ποτέ δεν το δώσαμε στην ελευθερία έκφρασης στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημιουργούς στο Ιράν το Ιράν το οποίο είναι στην επικαιρότητα με τις πυρηνικές απειλές, με τους κινδύνους ένοπλης σύραξης με το Ισραήλ, με την υποστήριξή του στον Μπασάρα Λασάντ κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή του κόσμου, να αναγνωρίσουμε, να στηρίξουμε ε, την προσπάθεια που κάνει η κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών στο Ιράν είναι πραγματικά τεράστια σημασία. Πρέπει να την αναγνωρίσουμε να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στους, στην πολιτική τάξη, ε, στους ηγέτες, στην κοινωνία και στη χώρα. Πρέπει λοιπόν ιδιαίτερα στην γυναίκα αυτή την Ιρανή να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα φέτος. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Στρίφλερ. Θα δώσω την προεδρία στην κυρία Τσίνισιν. E, drodzy koledzy, mm, po tych Λοιπόν, ακούσαμε την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων και θα προχωρήσει η συζήτηση στις υποψηφιότητες αυτές. Ε, στη συζήτηση μπορείτε όλοι οι συναδελφοί να πάρετε ε, μέρος. Έχουμε 40 με 45 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα είμαι αυστηρή λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ξεπεράσετε τα δύο με τρία λεπτά. Ποιος θέλει να πάρει μέρος λοιπόν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Προτασίεβιτς, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως ε, ακριβώς υπόθηκε, όλες οι αντιπροσωπείες αξίζουν της υποστήριξής μας. Αν μπορούσαμε <clears throat> να απονείμουμε πολλά βραβεία Ζαχάροφ θα ήταν καλό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλές χώρες όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται αντικείμενο σεβασμού, δεν υπάρχει ελευθερία τύπου, δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης και σχετικά με την υποψηφιότητα του κυρίου Μπαλιάτσκι, Μπιαλάτσκι συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή για να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιπροσωπεύει κινήματα τα οποία σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η φυλάκισή του η συνεχιζόμενη χωρίς ε, να έχει περάσει από δίκη προήλθε επίσης δυστυχώς από τα λάθη των εισαγγελιών δύο κρατών μελών. Ανάμεσα σε όλες τις υποψηφιότητες που αξίζουν τη στήριξή μας είναι ο κύριος Μπιαλάτσκι. Θυμηθείτε, ε, είναι στη φυλακή γιατί εμείς κάναμε λάθος. Είναι στη φυλακή γιατί έκανε λάθος ο Πολωνός και ο Λιθουανός εισαγγελέα ε, που τον εξέδωσαν. Συνεπώς λοιπόν αν δεν είχαν κάνει το λάθος αυτό δεν θα ήταν φυλακή. Πρέπει λοιπόν να τον τιμήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι τέσσερις ε, οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί είναι πραγματικά ε, άξιες. Έχω κάποια θέματα βέβαια με την ε, υποψηφιότητα από τη Ρουάντα. Δεν θέλω να προκαταλάβω την ουσία της συζήτησης, αλλά νομίζω ότι δεν έχει προετοιμαστεί η υποψηφιότητα αυτή με σωστό τρόπο. Αλλά αυτή είναι προσωπική μου γνώμη λόγω της γνώσης που έχω για τη συγκεκριμένη χώρα. Εμένω στην Ιρανική η υποψηφιότητα είναι η πιο τεκμηριωμένη, η πιο θα έλεγα τεκμηριωμένη και η πιο ενδεικνυόμενη στα πλαίσια της παρούσης διεθνούς συγκυρίας. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Σενισίν. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στον υποψήφιο τον οποίο πρότεινα. Κάποιες παρατηρήσεις μόνο για τη φύση αυτού του βραβείου το βραβείο αυτό, αν δούμε το τι έχει γίνει στο παρελθόν, δεν είναι μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε άλλα μέσα για να το mm. κάνουμε αυτό. Είναι μέσο για να θεσπίσουμε υψηλά επίπεδα προστασίας των θεμελιωδών αξιών και των ελευθεριών. Ανάμεσα σε αυτούς ε, οι οποίοι υποφέρουν, είναι πάρα πολλοί μάλλον αυτοί που υποφέρουν και δεν θα πρέπει εμείς να επιλέγουμε ανάλογα με το επίπεδο ταλαιπωρίας αν θέλετε, η απελπισία στο οποίο βιώνουν δυστυχώς εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Συν της άλλης, το βραβείο αυτό δεν θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια μιας κομματικής πειθαρχία, αλλά να είναι έκφραση των συναισθημάτων μας και των ιδεών μας για την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. E, nie widzę. Mm, e, Καλώς λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τα οποία παρουσίασαν τις υποψηφιότητές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη τα οποία πήραν μέρος στην συζήτηση και που ήταν παρόντες εδώ και υποστηρίζουν έναν κάποιους από τους υποψηφίους σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι κάτι το θα έλεγα πολύ συνηθισμένο. Ε, είναι μια ευκαιρία τα μέλη να γνωρίσουν ποιοι είναι οι υποψήφοι, να γνωρίσουν τι νόημα έχει το Φαβίο Σαχάροφ και τι <clears throat> σημασία έχει η ελευθερία του λόγου που δυστυχώς σε πολλές περιοχές του κόσμου τα τελευταία χρόνια υφίσταται επιθέσεις. Η ελευθερία του λόγου είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλες τις χώρες. Κόγκητο έργο σουμ. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Όταν αναφερόμαστε σε κάτι και σκεφτόμαστε σε κάτι πρέπει να μπορούμε να το πούμε. Το να αφαιρείτε το δικαίωμα έκφρασης, το να αφαιρείτε το δικαίωμα να συμμεριστεί κανείς τις ιδέες του με κάποιον άλλο, το να τον υποχρεώνει να υιοθετεί μια αυτό είναι κάτι που είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν γιατί ακούσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται να πούν τις απόψεις τους, για ανθρώπους οι οποίοι τολμούν να ομιλούν. Δεν συμφωνούμε σε αυτή τη φάση ένα συγκεκριμένο υποψήφιο, αλλά όλοι αξίζουν της υποστήριξής μας. Να σας πω ποια είναι τα επόμενα στάδια πλέον το αμέσως επόμενο θα είναι η ψηφοφορία για έναν μικρό κατάλογο, όπως λέγεται, τον συνοπτικό κατάλογο των τριών υποψηφίων θα γίνει με μυστική ψηφοφορία στις 9 Οκτωβρίου, τρίτη απογευματινή, σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης. Η διάσκεψη των Προέδρων στις 26 Οκτωβρίου θα πάρει την απόφαση ε, στο Στρασβούργο ο νικητής θα προσκληθεί στην κοινή συνάντηση των επιτροπών των αρμόδιων ε, στις 10 ε, ε, Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο θα δοθούν τα βραβεία την 12η Δεκεμβρίου, 12 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο και η Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου θα κάνει ό,τι το απαραίτητο για να προχωρήσουν οι ε, διαδικασίες. Ε,